Καλημέρα. Αρχίζουμε την ε, σημερινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη που εγκρίναμε χθε το πρωί. Ποιο είναι το επόμενο σημείο. Συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμός των Προτεραιοτήτων ω προ την πολιτική για το 2016. Ο κύριο Φερνάντο Ρούας είναι ο εισηγητή μα. Ε, θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. Και το σχέδιο σας το έχει στείλει μόνο στα αγγλικά, και προτιμώ τις τροπολογίες να τις εντάξετε στα αγγλικά και να τις στείλετε πριν την ε, Τετάρτη 27 ε, Ιουλίου ε, στη Γραμματεία. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα την ψηφίσουμε την έκθεση για 11 Οκτωβρίου είναι η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ πριν συνεδριάσουμε εμείς δηλαδή τον Οκτώβρη. Το Σεπτέμβρη πρέπει να, οπωσδήποτε να ψηφίσουμε, γι' αυτό σας πιέζουμε λίγο χρονικά. Και γι' αυτό θα είναι στα αγγλικά το σχέδιο έκθεση και γι' αυτό ζητάω τις τροπολογίες ε, στα αγγλικά για να προλάβουμε, αλλιώς δεν θα προλάβουμε να προετοιμάσουμε το σχέδιό μας. Είναι τεχνικές τώρα αυτές οι λεπτομέρειες ε, για το ρυθμό με τον οποίο θα εργαστούμε. Ο κύριος Ρούας τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για τη βοήθειά σας στη δουλειά που κάνω. Όλοι ξέρουν ε, ποιοι είναι οι περιορισμοί βάσει των οποίων λειτουργούμε εδώ και γι' αυτό έχω προετοιμάσει διάφορες τροπολογίες για να συμπληρώσω το κείμενο. Και λαμβάνοντας υπόψη αυτές τι τροπολογίες ε, παρουσιάζω την έκθεση. Ως προς την ε, πολιτική συνοχής, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπάρχουν συστάσεις για την Ευρωζώνη και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικέ αναχώρα συστάσεις, επιτρέποντας έτσι μεγάλη λεπίδραση, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς Ούτως ώστε να θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Μόνο έτσι θα σταθεροποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω σε σχέση με αυτό το ζήτημα ότι ε, εδώ και καιρό είναι χαμηλό το επίπεδο επενδύσεων ε, στην Ευρώπη και είναι αρνητική η ε, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σε ορισμένα κράτη-μέλη δυστυχώς όλος ιδιαιτέρως. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα ταχύτατα και με συνέπεια θα πρέπει να εφαρμοστούν τα επιχειρησιακά σχέδια καθώς και άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα που επίσης χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και καταθέτω μια σχετική τροπολογία τη σημασία του σχεδίου Juncker και την απαραίτητη γεωγραφική ισορροπία ούτως ώστε να ε, εξασφαλιστεί η προσθετικότητα και η συμπληρωματικότητα σε σχέση με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Συνέργειες επίσης ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία. Χτες εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι το συζητήσαμε αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει επανειλημμένα να τονίζουμε τη σημασία τους. Έτσι μπορούμε να επενδύσουμε με σύνεση τα χρήματα των φορολογουμένων και να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Με αυτές τις επενδύσεις, με το συνδυασμό των ταμείων, χρειαζόμαστε ισχυρές ε, δημόσιες αρχές ε, διαχείρισης και γι' αυτό ο βασικός στόχος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η ενίσχυση της πολυεπίπεδης ε, διαχείρισης και η δημόσια διαχείριση σε κάθετο σε οριζόντιο επίπεδο με εστίαση στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για τις κρατικές προμήθειες όλους ιδιαίτερως και για τον έλεγχο από πλευράς των πολιτών για αύξηση της διαφάνειας και καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε το συνδυασμό της πολιτικής συνοχής με το γενικότερο μακροοικονομικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε την ανάπτυξη με βάση τον κανόνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να υλοποιήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους στρατηγικής Ευρώπη 2020 και από αυτή την άποψη και θέλω να το τονίσω, είναι σημαντικό το άρθρο 164 της συνθήκης ε, της Λισαβόνας για την ε, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έτσι νομιμοποιείται η πολιτική συνοχή, διότι, η πολιτική συνοχή διότι καταγράφεται στις συνθήκες. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ε, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινού σχεδίου. Βάσει του άρθρου 157 τονώνεται η συνεργασία ανάμεσα στις ε, περιοχές, ε, στις πόλεις, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτή η αρχή λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας και λόγω κοντόφθαλμων οικονομικών επιχειρημάτων τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, η καλή οικονομική διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με σύνεση βάσει της προληπτικής αρχής και θα υπενθυμίσω ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους για να αποφευθούν κακές τοπικές επενδύσεις ε, ε, και να τονωθούν αυτές που χρειάζονται για την οικονομία των κρατών μελών, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βελτιστοποιώντας ε, τη δημιουργία θέσεων εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Για την εφαρμογή των μέτρων, στα πλαίσια της ε, διαδικασίας του 2016 και την επιβολή κυρώσεων στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, κάτι που αναλύει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να τοποθετηθώ προσωπικά. Είναι απολύτως άδικο, παράλογο οικονομικά και ε, μη πρόσφορο. Θεωρώ ότι είναι βαθιά αδικία αυτό που συμβαίνει στην ε, περίπτωση της Πορτογαλίας για την επιβολή των κυρώσεων, γιατί τιμωρείται και πάλι η χώρα, ενώ έχει καταβάλει τόσες προσπάθειες να επιστρέψει στην ανάπτυξη και μιλώ για τη χώρα, για τους πολίτες, για την κυβέρνηση, για τις επιχειρήσεις και υπενθυμίζω ότι έγιναν περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις, αυξήθηκε η φορολογία, μειώθηκαν κατακόρυφα οι δημόσιες δαπάνες. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος προσαρμογής και ε, ε, θα ήταν άδικο να γίνει ε, αυτή η εσπευσμένη κίνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό, αυτή η θέση βρίσκει τους σύμφωνους στην Πορτογαλία. Δεν υπακούει σε καμία οικονομική λογική. Αντίθετα με αυτό που ισχυρίζονται και εγώ θεωρώ ότι ε, δεν μας επιτρέπουν να αμυνθούμε. Πώς γίνεται τώρα αφού προσπαθούμε να επιστρέψουμε σε επενδύσεις, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να έχουμε παραγωγικές επενδύσεις, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, εκείνη την ίδια στιγμή να μας επιβάλλουν κυρώσεις. Το 2016 Χρειαζόμαστε υποστήριξη επενδύσεων, χρειαζόμαστε προγράμματα που έχουν εγκριθεί ήδη από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και χρειάζεται εφαρμογή του κοινοτικού πλαίσιου στήριξη, όχι κυρώσει. Όλη αυτή η διαδικασία που προανέφερε είναι περίεργη και ξαναλέω δεν αρμόζει από πολιτική σκοπιά να εφαρμοστεί και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη την γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη μετά το Brexit, μετά ε, την, ε, ε, τις πολιτικό μικροκομματικές εγκαταστάσεις ε, ε, ε, που δημιουργούνται σε διάφορες χώρες με τη δημιουργία ασταθών κυβερνήσεων με τη συμφωνία όπως, συμφων... όπως συζητούν κάποιου την υπογραφή νέων συνθήκων για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουν οι υπόλοιπες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την μακροοικονομική τροχιά που βρίσκεται η Πορτογαλία θα πρέπει να αποφευθούν ε, αυτές οι κυρώσεις ε, πάση θυσία. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές ε, δημόσιες δαπανές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι κάποια κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ θετικό που μπόρεσαν να λάβουν υπόψη αυτές τις συστάσεις στα επιχειρησιακού του σχέδια και έκαναν ειδικέ επενδύσεις, συγκεκριμένε επενδύσεις βάσει των εξάντε ρεσιμοτήτων. Και γι' αυτό ε, μέσα στην έκθεση μιλάω για τις ε, επενδύσεις των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, χάρη στις οποίες μπόρεσαν να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και μπόρεσαν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και ε, συμβάλαμε έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν θέλω και να αναφερθώ σε κάποιες ε, περιοχές ε, που πλήττονται από φυσικά μειονεκτήματα, έχουν πολύ ανίσχυρες οικονομίες, χρειάζονται λοιπόν ειδική υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Α, και τέλος, να μιλήσω για την στήριξη, για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα δηλαδή που ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να γίνεται σε εθελούσια βάση ε, η τεχνική αρρωγή στα πλαίσια τη πολιτικής συνοχής για τα διάφορα προγράμματα που γίνεται με πρωτοβουλία, ξαναλέω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο και δεν θα πρέπει να προδικάζει μελλοντικέ προτάσεις σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της ε, νομοδότησής σας, αλλά και για δήλωση, τη δήλωσή σας για την κατάσταση στην Πορτογαλία. Και τώρα θα πρότεινα να εστιάσουμε στην ε, γνωμοδότηση. Και θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις, ε, ξεκινώντας με τον κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο που είναι καλή βάση για το μέλλον, για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τις μελλοντικέ ε, προοπτικές. Ειδικά το σημείο 2, η προτάση που κάνατε, ε, ευθυγραμμίζεται με τις ε, δικές μας θέσεις. Έχουμε πρόβλημα εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και το συζητήσαμε χθες για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης πρέπει, όπως λέμε στα αγγλικά, go local, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σε επίπεδο πόλεων και περιοχών. Αυτά τα δύο σημεία λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στην έκθεσή σας. Ε, αυτά που λέτε για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, διότι θα πρέπει να επεκταθεί, θα πρέπει να μάθουμε ημένα από τους δε, να ανταλλάξουμε ε, τις βέλτιστες πρακτικές, ε, να δούμε από ποια προγράμματα έχει υποφεληθεί κάποια άλλη περιοχή. Όταν ήμασταν εμείς νέο κράτος μέλος, ε, στρέφαμε το βλέμμα μας στην Ουαλία, στη Σκοτία και μας βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το όφελος και μπορούμε να μάθουμε πολύ από συστήματα που λειτουργούν εύρυθμα σε τοπικό επίπεδο. Κάτι άλλο που επίσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι να τονίζουμε στην προγραμματική περίοδο πόση σημασία έχει η κοινωνική οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πώς ορίζεται η κοινωνική οικονομία, συνεργατική οικονομία, ενώσεις, σύλλογοι. Τέτοιου είδους οργανώσεις ε, μπορούν να έρθουν πολύ κοντά στους πολίτες. Έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Και όταν συζητούμε με φίλους από την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, εκεί βρίσκουμε και παραδείγματα και αποδείξεις πόσο σημαντική είναι η κοινωνική οικονομία για την κοινωνική συνοχή. Είναι σημαντικό που το αναφέρετε, λοιπόν. Και είναι εξίσου σημαντικό διότι ε, στις 7 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο αποφάσισε να την τονώσει αυτήν την κοινωνική οικονομία για να επιτύχει την ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Συμφώνησαν τα 28 κράτη-μέλη και ως αποτέλεσμα ε, υπάρχει ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προτείνει να καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία και αυτό να ενταχθεί στο, έγγραφο, στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και συμφωνούμε, είμαστε στο πλευρό του Συμβουλίου και της Επιτροπής για αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να προτείνω να το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Προσβλέπω στην καλή μας μελλοντική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γιουρέκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σχέδιο της είναι πολύ ισορροπημένο και εμείς έχουμε μεγάλες ανησυχίες από την άποψη του ECR για αυτό το θέμα και βεβαίως με λόγια το σύνολο του ECR και όχι για συγκεκριμένες αντιπροσωπείες, αλλά ήθελα να τονίσω δύο πράγματα στην έκθεση ω έχει αυτή τη στιγμή. Η Κοινέ και γενικέ διατάξει σε σχέση με το Ταμείο Συνοχή έχουν υιοθετηθεί στην προηγούμενη ε, θητεία και ίσως είναι η πιο επίμαχη η διατάξη για την διακυβέρνηση πλουρές κρατών μελών από τη στιγμή που για τα κράτη τα οποία βρίσκονται στην Ευρωζώνη και όντως η σχέση ε, με το Brexit και τις σχέσεις με την Ισπανία και την Πορτογαλία ε, Δεν φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγμή ε, να τα συζητήσουμε. Ε, τώρα, κοιτώντα τη συγκεκριμένη έκθεση, όπω και ο κύριο Ρούας, θέλουμε να εφαρμοστούν αυτέ οι διατάξει ε, ω ε, τελευταίο τελευταία επιλογή από πλευρά τη Κομισιόν. Εδώ λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλογικά με ισορροπημένο τρόπο και ότι κάθε πρόγραμμα, πρόταση αναστολή να χρησιμοποιηθεί όσο γίνεται λιγότερο. Θα πρέπει να είναι διαφανείς για διαδικασίες αλλά και επωφελής για τους στόχους ε, των, ε, της πολιτικής συνοχής και επίσης να υπογραμμίζουμε το θέμα ότι κάποιοι όροι κάποιες φορές χρειάζονται και είναι και ωφέλιμοι. Περνώντα τώρα στην παράγραφο 5 που αναφέρεται στο πρόγραμμα στήριξη των διευθυντικών αλλαγών, να τονίσω ότι το ECR μπορεί να στηρίξει τη δημιουργία αυτού του προγράμματο επί τη βάση του ότι χρησιμοποιείται ε, χρήματα από την τεχνική αρρωγή που ήδη υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο των ε, υφιστάμενων κονδυλίων δηλαδή. Ενώ εσεί μιλάτε για μεταφορέ από την τεχνική αρρωγή τη συνογή. Αλλά αυτό ε, θα πρέπει να το τονίσουμε, να χρησιμοποιούμε δηλαδή πολυστοχοθετημένα κονδύλια ή μη απορροφηθέντα κονδύλια. Τώρα η τεχνική αρρωγή βέβαια θα πρέπει να εξεταστεί λεπτομερέστερα. Αυτό είναι ένα γενικό σχεδιο που ισχύει για όλους τους τομείς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το διερευνήσουμε περισσότερο στους επόμενους μήνες εδώ της Επιτροπής μας. Πιο αποτελεσματική χρήση λοιπόν υποφιστάμενων κονδυλίων, απλοποίηση και μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου θα πρέπει να αποτελεί τη νέο κανόνα όταν ε, πρόκειται για χρηματοδότηση νέων αλλά και συνεχιζόμενων κυρωτικών δράσεων. Μπορεί να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες με βάση αυτές τις απόψεις στην πορεία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η από την Άλντε είμαι εγώ, οπότε να σας παρουσιάσω την γνώμη της Άλντε και θα τα πω όλα αυτά στα βουλγαρικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γούας για το... τη γνωμοδότησή του. Υπάρχουν συστάσεις αναχώρα που δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν να προωθήσουν την οικονομική ανάκαμψη και τις επενδύσεις. Υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι το πρόγραμμα που στηρίζει τις διευθυντικές αλλαγές θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο. Πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων για να έχουμε τον προπολογισμό που θέλουμε η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται πολύ αργά και γι' αυτό πρέπει να έχουμε maximum συμπληρωματικότητα και συνέργεια ανάμεσα στα διάφορα επενδυτικά ταμεία, τα διευθυντικά ταμεία και τα άλλα ε, χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως ε, τα μέσα ειδικών επενδύσεων ε, και τα υπόλοιπα. Θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 και να κάνουμε μία ε, έρευνα για την καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών των κονδυλίων ε, της Ένωσης σε σχέση με τους στόχους ε, Ευρώπη 2020. Η υπερχόμενη αναθεώρηση του πολιετούς ε, προγράμματος πλαισίου θα αυξήσει την προστεθέμενη αξία όλων των προσπαθειών και βέβαια συνδέεται αυτό και με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον στα μελη και γι' αυτό και οι συστάσεις αναχώρα καθώς και η αιρεσιμότητα εντός της πολιτικής ε, συνοχής ε, παίζουν ρόλο κλειδί διότι έτσι υπάρχουν σημαντικές πολιτικές επενδύσεις για, ε, επιρροές για το επενδυτικό περιβάλλον. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με αποτελεσματικό και υποθετικό τρόπο. Και κλείνοντας, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ασκήσουμε περισσότερες, να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες, δηλαδή εμείς και τα κρατη για την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών και την παραπληρηματικότητα των ε, χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογία στο σχέδιο χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Επόμενη η κυρία Ευχαριστώ. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή μας για την έκθεσή του. Δεν θα σας εκπλήξει, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και το έχουμε υπογραμμίσει. Δεν συμφωνούμε πάρα πολύ με το συνολικό βασικό ύφος της γνωμοδότησης, γιατί ως πολιτική ομάδα ανησυχούμε όλο και περισσότερο με την όλο και στενότερη σύνδεση και υποταγή της ε, ε, περιφερειακής ε, και διαστατικής πολιτικής στο βωμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συστάσεων αναχώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε τους στόχους πολιτικής συνοχής. Γιατί δημιουργήθηκε. Για να μειωθούν οι ανισότητες οι και οικονομικές μεταξύ των περιφερειών. Αυτή είναι η δουλειά τους και συχνά οι περιφέρειες δεν έχουν καν δικαίωμα συναπόφασης στις λεγόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τους ε, ε, φοράνε σαν κορσέι οι κυβερνήσεις. Ε, αυτό αφορά τις συστάσεις αναχώρα. Οι περιφέρειες όμως παρόλα αυτά είναι αρμόδιες για την υλοποίηση. Βεβαίω υπάρχουν συστάσεις αναχώρα που έχουν νόημα. Δεν θέλω καθόλου να το αμφισβητήσω αυτό, αλλά δεν ε, συμμεριζόμαστε το δικό σας ενθουσιασμό. Για παράδειγμα, εγώ δεν θέλω οι περικοπές των συντάξεων να θεωρηθούν εθάρρυνση ε, για ε, να μετατεθεί στην πολιτική συνοχή σε αυτό. Κατά τα άλλα, ο ίδιος ο εισηγητής έπεσε σε κάποιες αντιφάσεις με την γνωμοδότηση λέει θέλει να συνδέσει περισσότερο και ισχυρότερα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο την πολιτική συνοχή αφενό, αφετέρου διαμαρτύρεται για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην Πορτογαλία. Μα ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Έρχεστε στα λόγια μας. Γι' αυτό εμεί δεν θέλουμε να υποταχθεί η ε, πολιτική συνοχή στις απόλυτες επιταγές της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Και τέλος, δεν συμφωνούμε και πάρα πολύ με την πρόταση να υπάρχει νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με λεφτά πάλι από τη συνοχή. Κατά την άποψή μας αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο εξαίρεση, αν γίνεται να καταργηθεί και τελείως αυτή η δυνατότητα να παίρνουμε λεφτά από τη συνοχή για να τα δίνουμε εκεί. Και αντιστοίχως θα κάνουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ, επόμενος σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Ρούας. Ε, ε, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές οι προκλήσει και οι δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ξέρει τα οικονομικά ε, για οι προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα έχουν ε, υποχωρήσει. Τάτι. Δεν έχουμε και πολύ καλές στατιστικές για τη δημιουργία των ε, νέων θέσεων εργασίας. Τα οικονομικά λοιπόν είναι κάπως ζωφερά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγαίνει και λέει ότι επιβάλλει τώρα στην Πορτογαλία και την Ισπανία ε, τα όσα προβλέπονται για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Έτσι θα βοηθήσουμε τις χώρες, ε, παγώνοντας τη χρηματοδότηση, τα οικονομικά του στοιχεία. Παρακαλώ να μπει αυτό στην τελική γνωμοδότηση. Η πράσινη ε, ανέκαθεν ναι, φράζαμε εκφράζαμε επιφυλάξεις για τη χρήση αυτής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει η διαδικασία αυτή για τρεις χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις χώρα, πιστεύουμε ότι ο αριθμός τους θα πρέπει να μειωθεί. Ακόμα και αν βασίζονται στη καλή βούληση και σε συμπεράσματα πυρογνωμόνων. Ο αριθμός και μόνον όλων αυτών των συστάσεων χώρα καθιστά δύσκολη την εφαρμογή τους. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουμε τη στρατηγική του 2020, τους συγκεκριμένους στόχους. Παρ' όλα αυτά, Βλέπουμε να αυξάνεται η φτώχεια, δεν δημιουργούνται αρκετά γρήγορα νέες θέσεις εργασίας κτλ. Και η έκθεση δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η κρίση η ρωσική, η παγκόσμια κρίση στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση ορισμένων κρατών μελών. Θα ήθελα να συγχαρώ Ε, τον εισηγητή για τις επιφυλάξεις που εκφράζει ως προς το, το εάν η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει για να λυθεί η ανεργία. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που ο κόσμος μεταναστεύει, οι δικοί μας ξενιτεύονται. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θετικά βραχή πρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Εγώ βλέπω ολόκληρα χωριά και πόλεις να διάζουν, να ε, ρημάζουν ε, στη χώρα μου. Δεν, ε, δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να εγκατασταθεί εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μέτρα και πολιτικές που να εθαρρύνουν τον κόσμο να παραμένει στον τόπο του. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Νταμάτο. Ποιος θα πάρει το λόγο εξ ονόματος της ομάδας της. Ουδής. Δεν βλέπω κανέναν από την ομάδα της. Άλλη, η κυρία Μπρέσο. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα ακόμα μια φορά να εκφράσω τους προβληματισμούς μου, διευρύνοντας κάπως ε, την ε, λογική ε, για αυτό το θέμα. Εμείς βασικά έχουμε δύο μεγάλες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ε, πρωτότοκη, τη διαρθωτική πολιτική και τα διαρθωτικά ταμεία που σταδιακά θέλουν να δημιουργήσουν σύγκληση ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών παρεμβαίνοντας εις βάθος σε μικροοικονομικό στους τομείς που χρειάζονται εξυγχρονισμό αλλά και κυρίως επενδύσεις. Και μιλάμε βέβαια για διάφορες πολιτικές εκεί και παράπλευρα όπως είναι γνωστά έχουμε την γεωργική πολιτική και το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου που είναι κομμάτι των διευθυντικών ταμείων και παρεμβαίνουν για τις διευθυντικές αλλαγές στο γεωργικό τομέα και για τους άλλους τομείς παρεμβαίνουν τα διευθυντικά ταμεία με περίπλοκες παρεμβάσεις και στην αγορά εργασίας αλλά και στις κοινωνικές συμβολές που ε, καλύπτει το κοινωνικό ταμείο. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες πολιτικές και γι' αυτό και ο προγραμματισμός είναι επταετής και άρα πολιτικές που θέλουν να καλύψουν ανεπάρκειες ή δυσκολίες επενδύσεων σε διάφορους τομείς και παρεμβαίνουν με συγκεκριμένο τρόπο με αναπτυξιακές πολιτικές στην μικροοικονομία, στο σύστημα των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στη δημόσια διοίκηση για να στηρίξουν την οικονομία. Και μετά στη συνέχεια έχουμε την άλλη πολιτική που ενισχύθηκε στη διάρκεια της κρίσης με διάφορα μέσα. Έχουμε μια πολιτική που από χρόνο σε χρόνο και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Παρεμβαίνει λοιπόν αυτή η πολιτική με σωστό ή λάθος τρόπο, γιατί πολλοί συνάδελφοι και ο ίδιος ο ηγητής, θεωρούν ότι με λάθος τρόπο παρεμβαίνει και βεβαίως και έχουν γίνει και λάθη, αλλά και πολλές ε, ε, ε, προτάσεις ή συστάσεις από την άλλη πλευρά είναι σωστές, παρεμβαίνουν στους τομείς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ας πούμε, ζητά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, των συντάξεων, του κοινωνικού συστήματος και τα πρόνοιας κτλ. Αλλά δεν αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα και τις ανάγκες ε, της επενδυτικές του. Εξετάζει τη γενική λειτουργία της οικονομίας της χώρας, της εκάστοτε χώρας. Βεβαίως υπάρχουν εδώ διάφορα ζητήματα. Ε, ότι, ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα σε όλα αυτά ναι, ε, είναι συγκοινωνούντα ε, δοχεία και οι οικονομικές, οι μακροοικονομικές πρέπει να συνοδεύονται και από πιο στοχοθετημένε πολιτικές. Αλλά αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Εξάμενο είναι κάτι διαφορετικό. Προσπαθεί να συντονίσει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών και τους προπολογισμού τους και από την άλλη πλευρά να εντοπίσει να εντοπίσει ποιοι τομεί ή μάλλον ποιοι παραγωγικοί φορεί απαιτούν, χρειάζονται μάλλον αλλαγέ, μεταρρυθμίσει. Η απόπειρα που συχνά γίνεται να χρησιμοποιηθούν τα διευθυντικά ταμεία ώστε να επιτευχθούν και τα μακροοικονομικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το αυτό που κάνουν είναι να ζημιώσουν τελικά τα διορθωτικά ταμεία. Τα ζημιώνουν από την άποψη της χρησιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να πούμε ότι ναι, τα διορθωτικά ταμεία δεν κατάφεραν να, το εξή, να τροποποιήσουν τους μακροοικονομικού το φορείς, ε, μάλλον παράγοντε τη οικονομία. Μα δεν έχουν σχέση γιατί... Ε, και τα διευθυντικά ταμεία ε, άνθησαν όταν υπήρχε ούτως ή άλλως άνθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας χρειαζόμαστε άλλα μέσα, όπως το σχέδιο Juncker, που είναι ένα από αυτά τα μέσα. Έπειτα, το να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στα μέσα, τα επενδυτικά, μάλιστα, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά να χρησιμοποιείται η πολιτική σύγκλησης ε, ε, και συνοχής και ανταγωνιστικότητας των ε, διαφόρων ε, περιφερειών για να παρέμβουν στην στην μακροοικονομική πολιτική δεν είναι δική τους αρμοδιότητα και κινδυνεύουμε να κάνουμε μεγάλα λάθη και μπερδέματα διότι εάν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό που έχουν συμφωνήσει να κάνουν και κατά τη γνώμη μου για αυτή την πολιτική είναι κάτι διαφορετικό, όπως είπα, αλλά θέλουν να πάνε να τιμωρήσουν περιφέρειες και δαφικότητες που κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν, ε, αλλά αξιολογούνται με διαφορετικά κριτήρια, με διαφορετικά προγράμματα δεν πρέπει να, να εκριθούν με βάση το τι κάνουν τα κράτη και τις μακροοικονομικές πολιτικές που εμπίπτουν σε άλλα ε, σε αρμοδιότητες ε, εξάλλου. Όπως ξέρει και η Πρόεδρος, ε, γίνεται μια εις βάθος συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του εις πολιτική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εν γέννη και τη μακροοικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται εργασία πάνω σε, στην ιδέα ενός κώδικα σύγκλησης που θα ήταν πάλι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν θα είναι μεμονωμένε συμφωνίε που πάνω κάτω θα έχουν επιβληθεί. Γίνεται αντίθετα ένα μέσο πιο ευέλικτο με μεγαλύτερη δυνατότητα διαχείριση, καλύτερη διαχείριση, γιατί εκεί θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται παράμετροι κοινωνικού τύπου όπω αυτέ που είχαμε ζητήσει. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν στον εισηγητή μα ε, και ίσω και εγώ θα υποβάλω και κάποιε τροπολογίε κατά κάποιο τρόπο λοιπόν αυτό να το θυμίσει διότι όταν ε, ο εισηγητής διαμαρτύρεται για τη θέση και την επιβολή κανόνων στο μακροοικονομικό θέμα θα πρέπει ωστόσο να πούμε και ξεκάθαρα ότι είτε είναι δίκαιες είτε είναι, διά, ε, είναι άδικες ε, δεν θα πρέπει να αγγίζουν τα διευθυντικά ταμεία. Αυτή ήταν ανέκαθεν η θέση μας στην Περιφερειακή Επιτροπή η μακροοικονομική ερεσιμότητα στην ουσία έχει την τάση να συνενώνει τις δύο διαφορετικές πολιτικές. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την τάση στην Επιτροπή μας ανέκαθεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. Κύριος Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, είχα στην ΙΜΚΟ άλλη υποχρέωση. Μερικά σχόλια. Ήταν πάρα πολύ σαφής η τελευταία παρατήρηση. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Και η Ρέγγι το λέει ανέκαθεν αυτό, ότι δεν υπάρχει σχέση. Δεν είναι καλή ανάγνωση αυτή ε, των βημάτων που έχουμε θέσει. Και εγώ πιστεύω ότι βεβαίως υπάρχουν σχέσεις, αλλά πώς να το πω, μακροοικονομικά ε, είναι ένα θέμα και άλλο είναι τα μικροοικονομικά. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα. Ε, συστάσεις αναχώρα χώρα που μπορεί να τις εφαρμόσει και μπορεί και να μην τις εφαρμόσει. Έχετε έναν νέο που έχει σπουδάσει και δεν έχει δουλειά και έχει, ξέρω εγώ, 16 επιλογές. Ε, μπορείτε να του δώσετε και μια 17η πρωτοβουλία για το νέο δουλειά, δεν έχει ο άνθρωπος. <laughs> το σύστημα λοιπόν τη παιδεία ε, και τη εκπαίδευση είναι αυτό που χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ωραία αυτά που μας λέτε, οι πρασινάδες και οι διακλαδώσεις των συστάσεων. Αλλά ε, τι αποτέλεσμα έχουμε. τίποτα κλείνουμε τα μάτια, βάζουμε κάτω το κεφάλι και τρέχουμε να περάσουμε τον αυτοκινητόδρομο. Εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοιες σκέψεις και τέτοια συμπεράσματα. Και αν κοιτάξετε την έκθεσή μου, ε, ό,τι γνώμη και να έχετε για αυτήν, τα τρία τέταρτα του συστάσεων αναχώρα ε, αφορούν τη δική μας πολιτική. Ε, επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Και έρχομαι λίγο πιο κοντά τώρα στη διατύπωση του εισηγητή που λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, να έχουμε μέσα, εργαλεία και χρήματα, αλλά δεν ταυτίζονται πάντα οι στόχοι και οι πολιτικές των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έτσι κι αλλιώς οι επιτροπές νομοδοτούν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο λόγο στο τι θα γίνει, αλλά μπορούμε να συντονιζόμαστε, να συμφωνούμε. Όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους για τη συνοχή, για τις διαρθρωτικές πολιτικές Και σε ό,τι αφορά τώρα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δεν είναι του παρόντος. Αν καταφέρουμε εμείς να θέσουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων για τα μέτρα και τις συστάσεις ανά χώρα που πρέπει πραγματικά να εφαρμοστούν για να αποδώσουν, τότε θα έχουμε πετύχει. Για το 16.3 πρέπει να έχουμε μια ιδέα ε, λοιπόν τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς και πώς θα συνεργαστούμε. Στο, στην ίδια βάρκα είμαστε. Δεν είναι άλλη βάρκα η συνοχή και άλλη βάρκα τα οικονομικά, τα διαρθρωτικά. Μία είναι η βάρκα ευρωπαϊκή. Και δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε παράλυση η δική μας πολιτική γιατί θα την έχουν αποστραγγίσει. Αυτά έτσι ως κάποια σχόλια, κάποιοι προβληματισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εισηγητή για ε, το νέο αυτό πρόγραμμα στη γνωμοδότησή του, αυτό που προτείνει, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είχα την εντύπωση ε, από αυτά που άκουσα ότι Ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι μπορούμε να πάρουμε χρήματα από τη συνοχή για την ενίσχυση κάποιων μακροοικονομικών έργων και προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ισχύει. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο κατάφερε να διαπραγματευτεί να υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τεχνική βοήθεια και ένα κλάσμα αυτών των πόρων θα πάει στο νέο μέσο. Ένα κλάσμα επαναλαμβάνω για τεχνική βοήθεια και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εμπειρογνώμονες, ε, εθελοντικά όλα και κατόπιν συνεννοήσεως με τα κράτη-μέλη. Ε, διατίθενται λοιπόν εμπειρογνώμονες που μπορούν ενδεχομένως να βοηθήσουν για να δούμε πώς ε, εφαρμόζονται ορισμένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις των συστάσεων αναχώρα. Πώς τα λένε αυτά, country specific recommendations, το βρήκα. Λοιπόν, στις συστάσεις αναχώρα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή που το ξεκαθαρίζει. Δεν είναι αυτόματη η παράταση, είναι φάπαξ και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας και ούτε θα θεωρηθεί προηγούμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε στη γνωμοδότησή μας αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Are there any other? Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια ε, από τους συναδέλφους. Όχι. Ε, ε, έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ και ΡΕΤΖΙΟ. Ποιος θα πάρει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι σας. ΕΚΦΙΝ. No. Ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.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 για την πολιτική συνοχή. Δεν ξέρω ποιοι ήσασταν χτες παρόντες όταν ο Βάλτερ Δεφά μίλησε. Είναι δύο σημαντικά αυτά που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν σταθερή μακροοικονομική κατάσταση έτσι ώστε οι επενδύσεις να πιάνουν τόπο και να αποδίδουν. Στη νέα ε, πολιτική έχουμε εξάντε ε, αιρεσιμότητα για να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για την πολιτική ε, συνοχή, υπάρχει και η αναπτυξιακή και η επενδυτική. Για τις κυρώσεις και την πολιτική συνοχή, δεν θα μιλήσω για τις άλλες κυρώσεις που έχουν να κάνουν με τα μικροοικονομικά, γιατί αφορούν άλλη γενική διεύθυνση. Οι κυρώσεις περί των οποίων ομιλούμε αφορούν ε, υποχρεώσεις ανάληψη για το 2017 και όχι πληρωμές ενώ για το 14, 2015, 2016 έχουν ήδη καταβληθεί. Υπάρχουν κάποια ΕΣΠΑ που έχουν καθυστερήσει και τα είπε πολύ ε, ωραία χθες ο κ. Ντεφά ε, μέχρι τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κονδύλια να πιάσουν τόπο και να αποδώσουν ε, όσο γίνεται καλύτερα. Καθυστερήσει βεβαίω υπήρξαν. Για ποιο λόγο οι πληρωμές είναι στα σημερινά επίπεδα. Διότι η ανάληψη υποχρεώσεων έχει γίνει για τα τρία χρόνια και οι κυρώσεις δεν αφορούν τις πληρωμές, επαναλαμβάνω, και μόνο το 2017. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συζητούμε και σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα. Όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη, όπου χρειάζεται ε, να δίνουμε βοήθεια στους ανθρώπους που θέλουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα να προχωρήσει. Ευχαριστώ κύριος Ρούας. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύντομη παρέμβαση για να διευκρινίσω μια κατάσταση. Η αναφορά που έκανα στην κατάσταση των κυρώσεων ε, κατά της χώρας μου δεν έχουν σχέση με αυτή την έκθεση, αλλά θα καταλάβετε ότι κάποιος που παρακολούθησε μια συλλογική προσπάθεια ε, για να ξεπαράσουμε μόλις ε, κατά δύο δέκατα αυτό που απαιτούσε η Κομισιόν δεν καταλαβαίνω αυτήν την ε, προσέγγιση ε, σε αυτό το θέμα. Δεν ε, πιστεύουμε ότι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί όταν ακολουθεί το σωστό δρόμο και γι' αυτό και μόνο αναφέρθηκα σε αυτές τις κυρώσεις προς τη χώρα μου, κατά της χώρας μου που θεωρώ ότι είναι αντιπαραγωγικές γιατί δεν αλλάξαμε πορεία, είμαστε στον ίδιο και το σωστό δρόμο, το δρόμο που υπέδειξε η ίδια η Επιτροπή. Γι' αυτό ε, αναφέρθηκα σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα θα ήθελα να κάνω μια άλλη ε, ε, αναφορά και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, τις επικρίσεις τους, τα σχόλιά τους και φυσικά θα λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις. Δεν ήθελα να τονίσω κάτι ιδιαίτερα. Συνέλεξα όλες τα σχόλια και θα τα λάβω υπόψη. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη παρέμβαση που έχει να κάνει με την κοινωνική οικονομία και την πρόταση που έκανε ο συνάδελφος για προσέγγιση να ακούμε περισσότερο τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές. Τίποτα δεν με ευχαριστεί περισσότερο. Εγώ ήμουν πρόεδρος ε, ενό ε, Δήμου και ήμουν υπεύθυνο για το πρόσωπο των ε, τοπικών αρχών στις χώρες μου ε, και ε, το έχω αυτό το ζήτημα στην καρδιά μας. Και όπιτα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική είναι, είναι θεμελιώδη σημασία. Θα έλεγα ότι χάρη σε, αυτή, σε αυτές μπορέσαμε να αντέξουμε την κρίση και γι' αυτό και σας ευχαριστώ για την πρότασή σας που φυσικά και θα λάβω υπόψη. Ε, τώρα, σε σχέση με τις, ε, τη συνέχεια και τις ε, προσδοκίες που υπάρχουν ναι, φυσικά και θα δεχτώ τις απολογίες. σας. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους και την Επιτροπή, το σύνολο της Επιτροπής και ελπίζω ότι και στις συνεδριάσεις με τους κοιόδης εισηγητές θα είμαστε αποτελεσματικοί και με την ευκαιρία να σας ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές. Ευχαριστώ. σας ευχαριστούμε. Thank you. The, the whole meeting today will be... Ευχαριστώ. Ναι, όλοι οι συνεδρίαση σήμερα θα είναι σε, αυτές, ε, σε αυτό το κλίμα των ευχών. Yes, yes, yes, yes, yes. Σχόλια εκτός μικροφώνου. We can do this. We can do this. Okay. We, we, continue, we continue now Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο μας ε, σημείο, το θέμα της ε, ημερήσια διάταξη ε, που είναι ο Γενικός Υπερπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτος 2017, όλα τα τμήματα αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Η συγγητής μας είναι ο κύριος Βόν. Σήμερα ο κύριος Βόν μας υποβάλλει το σχέδιο γνωμοδότησής του και προτείνω την υποβολή των τροπολογιών μέχρι τις 22 Ιουλίου Παρασκευή το, στις 12 το μεσημέρι. Μπορούμε να ψηφίσουμε έτσι στις 8 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίασή μας γιατί η Επιτροπή Προπολογισμού θα ψηφίσει στις 11 Οκτωβρίου. Ε, αυτό ε, έχουμε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, το, η γνωμοδότηση The δεν θα είναι στο σύστημα, γι' αυτό ε, ε, θα καθυστερήσουμε. Προτείνω τι τροπολογίε να τι υποβάλλετε στα αγγλικά και να τις στέλνετε με email στην γραμματεία Reggie. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω και να δουλέψουμε βασικά ε, στα αγγλικά. Uh, uh, um, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω φυσικά το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει τώρα εκπονήσει το σχέδιο του προπολογισμού λίγο αργότερα από ό,τι ήθιστε φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, πάντως χαίρομαι που επιτέλους στόλαβα το σχέδιο. Οι συνάδελφοι σε αυτή την Επιτροπή θα γνωρίζουν ότι το εν τρίτο του προπολογισμού της Ένωσης στόχο έχει τη συνοχή. Και επίσης γνωρίζουμε πόσο σημαντικό επενδυτικό εργαλείο είναι η ε, εν λόγω πολιτική. Και σε κάποια κράτη-μέλη είναι το βασικό επενδυτικό εργαλείο για τα κράτη και τις περιφέρειες. Ο υπολογισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα κάθε χρόνο. Για το σχέδιο προπολογισμού του 2017 είχα ήδη εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με το 1β της ε, πιστώσης πληρωμών, τεράστια περικοπή, 27,3 δις, δηλαδή 23,5% κάτω σε σχέση με τον προπολογισμό του 2016. Τεράστια περικοπή για το 2017. στο, στην κατηγορία 1β. Ε, άρα λοιπόν και η ταχύτητα εφαρμογής θα πρέπει να επιταχυνθεί. Εν τω μεταξύ, εφόσον περισσότερα projects εγκρίνονται και αν δεν έχουμε τα χρήματα για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανελημμένες υποχρεώσεις, τότε θα καθυστερήσουν και οι πληρωμές στους δικαιούχους. Αυτή είναι η βασική μας ανησυχία. Όσοι ήσασταν εδώ εχθές και ακούσατε τον κύριο Ντεφά, είπε εκείνο ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα γιατί η περικοπή βασίζεται σε πληροφορίες που παίρνουν από τα κρατημέλη σε σχέση με την, το ρυθμό εφαρμογής και γι' αυτό εξήγησε η Κομισιόν ε, προτείνει αυτή την περικοπή 23,5% και φυσικά εμείς δεν έχουμε παρά να το πιστέψουμε. Ε, αλλά η Κομισιόν ίσως θα έπρεπε να κάνει μια κατανομή, μια ανάλυση των αναγκών των κρατών μελών για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια γιατί προτείνεται τόσο μεγάλη περικοπή. Επίσης θα είχα να πω ότι ως Επιτροπή θα έπρεπε να επιμείνουμε ώστε το Συμβούλιο να μην προβεί σε υπεραιτέρω περικοπές σε αυτό το νούμερο. Από ό,τι κατάλαβα χτες στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες για να αποκαταστήσουμε οποιασδήποτε περικοπές προτείνει το Συμβούλιο Βουλή στο σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής και ελπίζω πως και οι συνάδελφοι σήμερα θα το δεχτούν αυτό ως πρόταση. Πρόεδρε, εσείς μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα που είναι σύντομο και γρήγορο, αλλά ελπίζω πως οι συνάδελφοι θα διαβάσουν το σχέδιο, θα κάνουν τα σχόλια του σήμερα και θα καταθέσουν τις τροπολογίες τους εντός της προθεσμίας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους σκιώδες την σκιώδη συγγήτρια την κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιχαήλο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφό μας, συγητή για το έργο του και γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δύο σχόλια έχω να κάνω. It is evident that issue... Πρώτον, είναι προφανέ ότι το θέμα με τι καθυστερήσει πληρωμών και θα το βρούμε και πάλι μπροστά μα και θα μα εμποδίζει. Και μα έχει στοιχειώσει ξανά και ξανά. Την τελευταία φορά ε, ήμουνα εγώ στη θέση του κυρίου Βόνη, ήμουν συντάκτρια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πάλι. Από ό,τι φαίνεται, κάτι πάει στραβά έτσι, διαρθρωτικά στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά ταμεία και πώς δρομολογεί τις πληρωμές θα πρέπει να ανησυχήσουμε περισσότερο και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει μια αποτελεσματική λύση. Πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή χρειάζονται πηγόντως τα χρήματα. Δεν μπορούν να ε, ζήσουν είναι αυτή την αφόρητη καθυστέρηση πληρωμών. Για την απλοποίηση, μάλιστα, τα καταφέραμε και, και μάλλον τα χρειαζόμαστε και εμείς και οι δικαιούχοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως αντί να αναλωνόμαστε εδώ στην Επιτροπή με εκθέσεις που δεν είναι τόσο χρήσιμες και έχουν και περιορισμένη νομοθετική επίπτωση. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βον για την ρεαλιστική του προσέγγιση στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς. Thank you very much, President. Ευχαριστώ την έκθεση και τις προσπάθειες που γίνονται για την ε, επικέντρωση επί των αποτελεσμάτων για τον προϋπολογισμό και καλούμε την Επιτροπή να πλουστεύσει περισσότερο την διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα δεν βάσει στον τίτλο 1β τα κονδύλια δεν επαρκούν για τις ε, πιστώσεις ανάληψης επιπληρωμών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, εγκαίρως να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τη συμβολή του στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Επίσης, διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στο 1β του σχεδίου προϋπολογισμού το 2017 ανάμεσα στις πιστώσεις άλλων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληροφοριών. Ε, περάσαμε στα 17 δισεκατομμύρια από 16,3 και το 2017 θα αυξηθούν περισσότερο οι πιστώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυξημένους πόρους. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις πιστώσεις πληρωμών. Θα υπάρχει αρνητική επίπτωση στο backlog, αυτές τις καθυστερούμενες πληρωμές και θα συσσωρευτούν τα πλήρωτα τιμολόγια στο δεύτερο, στη δεύτερη περίοδο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε. Εγώ είμαι η επόμενη σχεώδης για τους φιλελεύθερους. Ναι. Και θα τα πω στη μετρική μου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, για αυτή την τόσο θετική προσέγγιση που διαπιστώνω μέσα στο σχέδιο έκθεσης. Όμως έχουν περικοπεί ε, σοβαρά τα κονδύλια για τη συνοχή. Για το 2000, ε, από σχέση με το 2016 είναι μια μείωση 20,3% όπως είπε ο ε, και ανησυχώ ιδιαίτερα. Όμως, ε, για την απορρόφηση του χρόνου από των επενδυτικών και διαρθρωτικών ταμείων μπορούμε να αναμείνουμε ε, την επίτευξη του ανωτάτου επίπεδου δεδομένων των προγραμμάτων που τρέχουν και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουμε αυξημένες πιστώσεις, ε, όχι μειωμένες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα κατάλληλα κονδυλία για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που υπάρχουν ήδη για να μπορέσουν να καλυφθούν οι πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2017. Για να μην υπάρχουν καθυστερούμενες ε, και πληρωμές και δεδουλευμένοι τόκοι που πρέπει να καταβληθούν. Εάν δεν εφαρμοστούν τα προγράμματα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ε, θα υπονομευθούν οι στόχοι της ε, Ευρώπης 2020, ε, της πολιτικής συνοχής, θα πληγεί η ίδια η εξοπιστία της πολιτικής. Μόνο με την εκπλήρωση αυτής της πολιτικής θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσει των κρατών μελών θα έπρεπε να αποτιμήσουν ε, ο, σε ένα ενδιάμεσο στάδιο τα αποτελέσματα όλων των προγραμμάτων και αν διαπιστωθούν ελλείψεις θα, θα πρέπει να υπάρξει θεώρηση. Εάν δεν υπάρξει διόρθωση τότε θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις πιστώσεις σε άλλα προγράμματα που πληρούν τα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργεί σε διάδραση με τα κράτη-μέλη όταν ζητούν τροποποίηση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων με στόχο να υπάρχει ένας καλύτερος συνδυασμός των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και των ταμείων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων όπως του προσφυγικού. Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους ταμείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να κατοχυρώσουμε και η διασταυρούμενη χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Τελικά, τι είναι σημαντικό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να απορροφούν το σύνολο των κονδυλίων από όλε τι δυνατέ πηγές και ε, φυσικά τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Ε, εξασφαλίστε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ε, των επενδύσεων που γίνονται βάσει του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο και ε, ε, αντί για την κυρία Βάρνα, θα μιλήσει ο κύριο Δρόπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Μόνικα Βάνα. Ζητά συγγνώμη που σήμερα δεν μπορούσε να παρευρεθεί η συνεδρίαση. Εκφράστη την ευγνωμοσύνη της για την καλή δουλειά που γίνει για αυτή την έκθεση και έχει διάφορες ε, προτάσεις. Μέσα στην έκθεση μιλάμε για την ε, περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ως προς τη στρατηγική 2020 και η απλούστευση θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τη στρατηγική. Τονίζεται η σημασία της ε, πολιτικής συνοχής και κατονομάζονται τα πραγματικά προβλήματα που οφείλονται στις ε, καθυστερούμενες πληρωμές. Τα ε, εθνικά κονδύλια θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει των ε, νέων στατιστικών ε, στοιχείων στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρο ε, θα πρέπει να επικρατήσει η αλληλεγγύη και σε άλλες χώρες όπως η Τσεχία, η Κροατία, η Σλοβενία θα ζητήσουμε επιπρόσθετη στήριξη για τη δημιουργία προσθέμενης αξίας, ε, ε, ανεργία των νέων, προσφυγικό, μεταναστευτικό, θέλουμε να είναι πιο δυναμικά τα μέτρα επίσης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Προτείνεται το 20% είναι δεν είναι αρκετά φιλοδοξό ο στόχος στα πλαίσια των ε, ε, ε, υποχρεώσεών μας της COP21. Η ενσωμάτωση επίση τη ε, διάστασης του ισότητα των δύο φίλων είναι κάτι που δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε στη στρατηγική μας. Ευχαριστούμε. Thank you. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Μανίστερόι και μετά ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ επίσης για ε, την εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση και το κείμενο. Μήπως θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με την πρόταση που υιοθετήσαμε στο ψήφισμά μας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που λέγουμε το εξής. There, should not be any... Δεν θα πρέπει να επιστρέφονται χρήματα στα κράτη-μέλη όταν δεν ε, δαπανώνται τα κονδύλια με συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο. Ε, υπάρχει ένα κείμενο που το ψηφίσαμε και το εγκρίναμε. Ε, στην έκθεση για την ενδιάμεση αναθεώρηση θα μπορούσαμε να το βάλουμε και εδώ. Γιατί έχουμε ένα ορίζοντα πολιτή. Και αργότερα αυτό θα συσσωρεύσει οι περίμερες πληρωμές. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσουν εκατομμύρια ε, στους καθαρούς συνεισφορείς και μετά να λέμε έχουμε προβλήματα στις γιατί τους γύρισαμε τα λεφτά. Γιατί ε, αφορά εμάς αυτή η υπόθεση, την Επιτροπή μας, την ανάληψη υποχρεώσεων ε, που θα έχουμε στο προσεχές μέλλον και τα καθυστερούμενα το backlog που θα βρούμε μπροστά μας επίσης τα επόμενα έτη. Παρακαλώ κοιτάξτε αυτή την τροπολογία και αν μπορεί ο εισηγητής να το υιοθετήσει, δεν χρειάζεται να το καταθέσουμε. Είστε πρόθυμος να πάρετε αυτό το κομμάτι από το ψήφισμα, ε, από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Oh, Α, συγγνώμη, δεν σας είδα κύριε Βούτα. Προηγουμένως είπα ότι είστε επόμενος ομιλητής, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είμαι και εγώ εισηγητής, ξέρετε, ε, και σκιώδης ε, για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την προσοχή σε ένα κίνδυνο που έχουμε ενώπιον μας και ελοχεύει. 23,5% μειώνονται τα διαρθωτικά ταμεία. Κάπου υπάρχει ένα λογικό σφάλμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε συζητήσαμε για τα πλεονεκτήματα της πολιτικής συνοχής σε όλα τα κράτη-μέλη. Και σε χώρες που ζουν από τα διαρθωτικά ταμεία. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που επωφελούνται και οι πάντες είναι ικανοποιημένοι. Τώρα αυτό είναι κατανόητο. Γιατί πρέπει να περικοπούν κατά 23,5% ακριβώς αυτά τα ταμεία. Υπάρχει μια τέτοια τάση η Φέρπουσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώνει τα κονδύλια της συνοχής και της κοινή γεωργικής πολιτικής κατά τα άλλα. Ε, να μιλάς μετά για περισσότερη Ευρώπη όταν συνέχεια έχουμε περικοπές σε αυτά τα κονδύλια. Εκεί ζει ο κόσμος στην Ευρώπη και δεν στο πετσί του, σε αυτές τις πολιτικές. Όταν έχουμε και θετικέ συνέπειε και τις βλέπει ο πολίτης. Ευχαριστώ. Άλλο. No, I'll give the floor uh, θα δώσω το λόγο τώρα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, ε, έτσι δεν Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Φιλίπ Ζωή. Ασχολούμαι με την ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στη DG Regio. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, ε, κατανοώ τις ανησυχίες σας και τώρα θα προσπαθήσω να εξηγήσω ε, πώς καταλήξαμε σε αυτά τα ποσά του σχεδίου προϋπολογισμού 2017. Για το 2017 ε, έχω να πω ότι είναι μεταβατική χρονιά. Γιατί, διότι για τα παλιά προγράμματα 2007-2013 υπάρχει μεγάλη μείωση και ταυτόχρονα μεγάλη αύξηση για τα νέα προγράμματα. 33% αύξηση για τα νέα προγράμματα. Για το 2007-2013 είναι μείωση για τα παλιά προγράμματα και φέτος θα πληρώσουμε τους τελευταίους λογαριασμούς βάσει των προβλέψεων των κρατών μελών ε, δεν θα, θα εκλείψει το backlog δηλαδή εκτός από τα προγράμματα που υπάρχει παράταση και του χρόνου θα αρχίσουμε το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013. Η προθεσμία για την υποβολή των ε, παραστατικών για να κλείσουν τα προγράμματα γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκπνέει το Μάρτιο 2017. Ε, το 17 όμως δεν θα κλείσουν ε, τα περισσότερα προγράμματα, το 18 ή το 19 θα κλείσουν. Για τα προγράμματα 2007-2013 είναι περιορισμένα τα κονδύλια για το κλείσιμο, γιατί είπα δεν θα γίνει το 2017. Είμαστε όμως πιο αισιόδοξοι σε σχέση με αυτά που είχαμε προβλέψει το 2010. Θα κλείσουν ταχύτερα τα προγράμματα, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Για πάμε τώρα στα νέα προγράμματα, 14-20. Οι πιστώσεις, είπαμε, αυξάνονται κατά 32-33% από την ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ρέτζιο. Κάνουμε τις προβλέψεις μας ε, βάσει του μοντέλου πληρωμών της προηγούμενης περίοδου. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της νέας προγραμματικής περίοδου και κάνουμε διασταυρούμενους ελέγχους, όπως είπε και ο κύριος ε, Νταφάχτες. Κάνουμε τους διασταυρούμενους ελέγχους λοιπόν βάσει των προβλέψεων των κρατών μελών που μας υπέβαλαν πέρσι τον Ιανουάριο. Είμαστε ελαφρώς ε, πίσω από τις προβλέψεις των κρατών μελών. Γιατί, διότι ε, υπάρχει υπερεκτίμηση από πλευρά τους στις προβλέψεις τους, αυτό το ξέρουμε από την εμπειρία μας. Ε, όμως, ε, ως επιτοπλίστων ευθυγραμμιζόμαστε με τις προβλέψεις τους. Ο προϋπολογισμός επιτρέπει λοιπόν αυξήσεις για τις αποζημιώσεις, ε, για τις ε, πληρωμές για τα νέα προγράμματα Ξέραμε, ξέρουμε φυσικά ότι υπήρχαν προβλήματα στις πληρωμές την προηγούμενη περίοδο και ξέρουμε ότι δεν πρέπει να περικοπούν οι πιστώσεις πληρωμών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δύο παρατηρήσεις ζητάει ο συγητής προβλέψεις. Τα δώσαμε αυτά το Φεβρουάριο στις εσωτερικές συσκέψεις για τις πληρωμές. Θα σας ξαναδώσουμε τις πληροφορίες όμως και θα σας εξηγήσουμε πώς ακριβώς ε, συνδυάζουμε τις προβλέψεις με τις πιστώσεις. Και δεύτερο το θέμα του backlog. Για τα νέα προγράμματα, για τις καθυστερήσεις πληρωμών που ε, προβλέπονται. Στο πολυεδέστημα νομικό πλαίσιο υπάρχει ένα εργαλείο αποφασιστική σημασία για αυτή την περίοδο. Δεν το διαθέταμε στο παρελθόν. Το Global Margin for Payments, το συνολικό περιθώριο για τι πληρωμέ. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει στο πολιετές να μεταφέρουμε τις πιστώσεις από τη μία χρονιά στην άλλη. Και είναι πολύ σημαντικό διότι μας επιτρέπει να εξομαλύνουμε το προφίλ των πληρωμών, μεταφέροντάς τες από τη μία χρονιά στην άλλη, εκπληρώνοντας τις ανάγκες της πολιτικής συνεχής, ούτως ώστε τις πιστώσεις να τις έχουμε όταν ε, ε, στέλνουν τα κράτη-μέλη τα αιτήματα προς Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. κύριος Βον θέλει να κάνει τις καταληκτικές σου παρατηρήσεις. Ναι, ναι. Ευχαριστώ για τα σχόλια, για το μεγάλο φάσμα ζητημάτων και κάποια νέα ζητήματα από κάποια σημαντικά. Ε, γιατί έχουμε και το προσφυγικό, την απενεργία των ε, την, το θέμα της απλούστευσης, ε, το θέμα των εθνικών κονδυλίων, ο Λάμπερτ μας είπε να μην επιστραφούν στα κράτη-μέλη τα κονδύλια που δεν έχουμε απορροφήσει, που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Θα το δούμε σε σχέση με την πρότασή του. Ε, η βασική εστίαση ήταν ε, ε, στο, για το, στο 1β για το 2017 και την μείωση 23,3% και τον backlog των πληρωμών οι καθυστερούμενες πληρωμές 2 δις προβλέπονται για το τέλος του 16 αλλά φαίνεται ότι θα αυξηθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί τις επόμενες χρονιές. Να μας ξαναστείλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Προβλέψη των Κρατών Μελών για να το δούμε. Ε, θέλουμε μια διευκρίνηση από πλευράς Επιτροπής ε, και, και για τη μείωση του 23,5%. Θέλουμε να το μελετήσουμε το θέμα. Για την πρόταση η υποστήριξη των τροπολογιών από ή από μένα για αποκατάσταση των περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο ελπίζω να είναι μια πρόταση που θα δεχτούν οι συνάδελφοι. Θα καταθέσω ειδική τροπολογία για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πέρα τη συζήτηση. Συνεχίζουμε. Ε, Παρουσίαση ε, του σχεδίου έκθεσης ιδίω πρωτοβουλία του κ. Τσίκο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύη. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα που έχουμε για να καταρτήσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύη. Μικρός Τσίκο. Στι 24 Μαου παρουσίασε το σχέδιο έκθεση. Οι συναρμόδιες επιτροπές, όπως η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ε, θα ψηφίσουν τη δική τους έκθεση, ίσως και να την έχουν ήδη ψηφίσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εμείς πάντως τον Οκτώβριο μάλλον θα ψηφίσουμε ε, για τις τροπολογίες 12 το μεσημέρι 19 Ιούλιο, Τρίτη. Εντάξει, κύριε Τσίκο. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω γνωρίζουμε, συνάδελφοι, τον Οκτώβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση για τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2014. Η έκθεση παρουσιάζει μια, την ιδιαίτερη καυτή κατάσταση και πιστεύω πως είναι μια ευκαιρία για να εξετάσουμε την λειτουργία αυτού του μέσου αλληλεγγύης η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε να, να, να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλία. Όπως υπογραμμίσατε, είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς όλες τις επίγουσες καταστάσεις και τις ε, καταστροφές. Ε, όμως οφείλουμε και είναι δυνατόν να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνεπειών τους. Στην διαχείριση των, των φυσικών καταστροφών ε, και των θεομηνιών υπάρχουν πάντοτε διάφορες φάσεις. Ε, πρώτη είναι η διαπίστωση ε, της δύναμης της φύσης που συνοδεύεται από, μια... από το δέος και καλύπτεται από τις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες βοήθειας. Ε, Όμω εμεί θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για τη δεύτερη και την τρίτη φάση, γιατί μετά από την διαχείριση τη άμεση ε, πήγουσα ανάγκη, τα θύματα πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, την διόρθωση των ζημιών, που πρέπει να είναι βιώσιμη. Κάποιε πτυχέ τη διαχείριση του Ταμείου Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπιστούν και θα θέλαμε να τονίσουμε τη ταχύτητα παρέμβαση, που είναι και καθώ και σε μια απαραίτητη πολιτική πρόληψη που συμβαδίζει με την συμπληρωματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης και άλλων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό και μάλλον πιο συγκεκριμένα της πολιτικής συνοχής. Ο εισηγητής θέλει να τονίσει τη συνεργασία που θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ανάμεσα στο εθνικό επίπεδο και τις τοπικές ή ε, περιφερειακές αρχές. Αρχίζω με την ταχύτητα της αντίδρασης. Ε, λόγω της του πρόβλεπτου χαρακτήρα της, μια φυσική καταστροφή όχι μόνο ε, αφήνει άναυδους τους πληθυσμού που έχουν ε, πληγεί, αλλά και τις δημόσιες αρχές που πρέπει ξαφνικά να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες δαπάνες. Από την αρχή της δημιουργίας αυτού του ταμείου, ο νομοθέτης προέβλεψε ένα συγκεκριμένο όρο ε, προθεσμία 10 εβδομάδων για την υποβολή ε, των ετοιμάτων. Αυτό θα έπρεπε να επιτρέψει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Όμως, στις πρώτες ε, χρονιές λειτουργίας του Ταμείου έδειξαν ότι πρόκειται για μια περίοδο εξαιρετικά σύντομη. Ε, στην αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας το 2014 η προθεσμία για την υποβολή ετοιμάτων επεκτάθηκε στις 12 εβδομάδες. Αυτό δεν προχωρά προς την κατεύθυνση του αιτήματο του εισηγητή, όμως οι τοπικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε το χρόνο να προετοιμάσουν τα σφακέλους και να ε, καθυστερήσουν περισσότερο. Γι' αυτό και αυτή η παράταση δεν είναι αντιφατική γιατί έτσι οι τοπικές αρχές μπορούν καλύτερα να προετοιμάσουν ε, του φάκελου τους που θέλουν υποβάλλον. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η ταχύτητα επεξεργασίας των φακέλων είναι πολύ σημαντική από τη στιγμή της υποβολής του πλήρους ε, φακέλου στις 12 εβδομάδες. Όλα τα επίπεδα λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να λειτουργήσουν ε, αποτελεσματικά τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο των υπηρεσιών της Κομισιόν ώστε τα χρήματα να, απελευθερωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τα θύματα δεν πρέπει να αισθανθούν ότι έχουν ε, εγκαταληφθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι επίγον επίγουσα η έκκληση αφορά τις μεγάλες ε, φυσικές καταστροφές που έπληξαν ε, τις χώρες του Νότου ε, που ούτε ούσοι είχαν αποδυναμωθεί λόγω της κρίσης και αναφέρομαι στη γη μου, στη, στη Σαρδινία όπου μετά από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2013 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.700 πλήγησαν σε πολύ σοβαρό βαθμό. Οι υπηρεσίες βοήθειας που παρεμβαίνουν αμέσως μπορούν να, κάπως να περιορίσουν τι αρνητικές επιπτώσει τη φυσική αυτή καταστροφή τη Ομινίας. Όμω ο νομοθέτη ακριβώ πρέπει να στηρίξει την αλλαγή των διαδικασιών ώστε να είναι πιο προσαρμοσμένε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να αποφευθούν περιπτώσει όπω αυτή της κρατίας του 2013 όπου δόθηκε η σύμφωνη γνώμη 17 μήνε μετά την κατάθεση του αιτήματο. Όταν είναι επίγουσα η κατάσταση πρέπει να είναι επίγουσα και ανταπόκριση. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση 1,5 χρόνο πέρασε πριν να φτάσουν τα χρήματα στους ε, πληγέντες. την το άλλο μεγάλο θέμα για την πρόληψη, εκτός από την πρόληψη, είναι η συμπληρωματικότητα, παραπληρωματικότητα. Πολύ συχνά, πολύ αργά μετά από μια θεομηνία φτάνει η φάση της πρόληψης, ενώ θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο τμήμα και άμεσο. Η αποκατάσταση των έργων που έχουν καταστραφεί ή οι διορθώσεις σε υποδομές επισκευέ σε υποδομές ε, θα πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπουν τα πράγματα ξανά στη φυσιολογική του ε, ροή. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει παραπληρωματικότητα ανάμεσα στο Ταμείο και στο Ταμείο Συνοχή. Και έπειτα υπάρχει και το μεγάλο θέμα τη διαφάνεια, επί το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε μάλλον, ε, αλλά είμαστε ήδη σε εξαιρετικό επίπεδο και έχουμε την συνεργασία ανάμεσα στα επίπεδα Λήψη αποφάσεων. Πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ε, στη διαχείριση του Ταμείου, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κονδύλια που δίνονται ως αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από μια φυσική καταστροφή θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στη, στα επίπεδα λήψης αποφάσεων και η συνεργασία επίσης ανάμεσα στις ε, αρχές που πρέπει να αποφασίσουν. Αυτό δεν αμφισβητείται, ωστόσο θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή στις μηχανισμούς συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και ε, στις τοπικές αρχές σε επίπεδο κάθε κράτο μέλους. Επίσης, συστήνουμε καλύτερη επικοινωνία με το κοινό στη διάρκεια όλη τη διαδικασία. γιατί έτσι οι δικαιούχοι ή ενδιαφερόμενοι να μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα τη διαδικασία για κάθε αίτημα. Ε, αυτό θα μπορούσε να διοργανωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την προπόθεση ότι θα θεσπιστεί μια ένα συγκεκριμένο ρούζι των πληροφοριών. Τέλος, πιστεύω ότι η εργασία και η συμβολή των συναδέλφων και στην προηγούμενη φάση ήταν πολύ σημαντική πολύ σημαντική και πολύ συγκεκριμένη, αλλά πιστεύω ακόμη περισσότερο πως στην, στην φάση των τροπολογιών θα μπορέσουμε πάλι να υπογραμμίσουμε και να ε, διευκρινίσουμε κάποιες στοιχές, όπως αυτό που μου είναι ιδιαίτερα αγαπητό, είναι το θέμα της, αποφάσης... της, της ε, ταχύτητας, της επιτάχυνσης μάλλον, γιατί ε, ο, αυτοί που σήμερα παίρνουν, μάλλον αυτοί που σήμερα πέφτουν θύματα μιας καταστροφής ε, σε σχέση με την κατάστασή τους ε, και παίρνουν τα χρήματα μετά από ένα, ένα, μισή χρόνο, αυτό είναι μια ζημιά μετά αναπότρεπτα που δεν μπορεί να αντιστραφεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Ε, η δραστηριότητά του και η ζωή του έχει ήδη καταστραφεί. Και γι' αυτό θα προτείνω με συγκεκριμένε τροπολογίε, συγκεκριμένε δράσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη. Η κυρία Κρέλ, εξ του κυρίου Πίτσουλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σκιώδη ηγητή μα δυστυχώ κολλείται και με, με παρακάλεσε να σα διαβάσω όσα θέλει να πει και θα τα διαβάσω στα αγγλικά. Ε, κύριε Σπίτσουλα, ευχαριστεί τον εισηγητή για το έργο του και την έκθεσή του από τη δημιουργία του μέχρι το περσινό Ιούλιο έδωσε το Ταμείο 3,8 δις ε, μετά από 69 αιτήματα από 24 κράτη-μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από επανειλημμένες απόπειρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τελικά εγκρίθηκαν το 2014 κάποιες διατάξεις για αλλαγές των κανόνων. Εγκρίθηκαν προκαταβολές και επίσης οι χώρες δικαιούχοι έχουν περισσότερο χρόνο να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια αυτή. Και ε, ε, διευκρινίστηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των θεομηνιών. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία των πληρωμών των εγκεκριμένων κονδυλίων παραμένει αργή. Ακόμα και μετά τη μεταρρύθμιση χρειάζεται τουλάχιστον 8 με 10 εβδομάδες και στην πράξη πολύ περισσότερο 6 με 8 μήνες. Θα πρέπει ενδεχομένω να κοιτάξουμε μήπως ε, αυξήσουμε τους πόρους έτσι ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε ε, περισσότερη ζημιά αυτή τη στιγμή ότι μόνο το 3 με 5%. Επίσης, ζητούμε πλήρη διαφάνεια στην δαπάνηση των κονδυλίων εντός της προθεσμίας που τίθεται. Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν μιλάει για το κατόφλι ε, των θεομηνιών να είναι στο 1% του ΑΕΠ και κάτω. Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση αυτή θα πρέπει να ε, δίνει και παραδείγματα επιτυχή και αποτυχημένα ε, σε σχέση με την εποχή που ιδρύθηκε το Ταμείο Αυτοαλληλεγγύης να έχει μεγαλύτερο όραμα και προοπτική για το μέλλον σε σχέση με το 14 που συστήθηκε. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση θα πρέπει να ε, αποσυνδεθεί γιατί υπάρχουν διαφορετικά ταμεία. Το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, έχει να κάνει με θεομηνίες και όχι με πρόσφυγες. Θα κάνω και δραπολογίες και χαίρομαι για τη μελλοντική μας συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Και συμφωνώ με όλες αυτές τις ευχές για καλές διακοπές. Γιατί και αυτή ήταν η τελευταία μου δράση εδώ πριν τις διακοπές. Να ξεκουραστείτε. Κατά τα άλλα, Πορτογαλία θα πάω. Τέλη Αυγούστου για να υποστηρίξω και τον κύριο Γουάς. Okay, thank you. Thank you for the good... Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας. Ε, δεν βλέπω τον κύριο Ποέβα, δεν πειράζει. Ο κύριος Μίλτενμπεργκ, σκιώδη ηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πραγματικά πολύτιμη η έκθεσή του. Συμφωνούμε για την τελευταία αναθεώρηση ε, των κανόνων του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 2014 έχει γίνει η προηγούμενη και τώρα είναι πολύ νωρίς για να προτείνουμε και νέα. Ε, συμφωνώ γενικά με τον εισηγητή, αλλά να τονίσω τρία ε, θέματα. Πρώτον, η ταχύτητα με την οποία κινητοποιείται, η σημασία της πρόληψης και ε, η υποστήριξη για τις αμυνίες. Πρώτον, η ταχύτητα βεβαίως θα πρέπει να μεγαλώσει. γρήγορα να εγκρίνονται, αλλά γρήγορα και να εκταμιεύονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει το συντομότερο, είναι επίγουσα αυτή όταν ζητούν να κινητοποιηθεί. Τώρα αυτές οι ολιγορίες και οι διαφυταλαντεύσεις και από τον Άννα στον Καγιάφα, ε, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, τι νόημα έχει. Είναι επίγουσες οι καταστάσεις και είναι οι ζωές των πολιτών. Δεύτερον, σωστά μιλάει ο για τη σημασία της πρόληψης. Θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή Ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή ε, αυξάνονται οι κίνδυνοι των θεομηνιών. 8 δισεκατομμύρια προβλέπονται για την πρόληψη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καινοτομία ε, και να ενισχύονται τέτοια έργα. Για να μειώνονται όχι μόνο τα δεινά του ανθρώπου, αλλά και γενικότερα ε, της φύσης. Τρίτον, στο 14, παράγραφο 14 λέει ο συγητής ότι στις θεομηνίες η ενίσχυση θα πρέπει να είναι στο 1% του ΕΠ της σε λόγω περιφέρειας. Εδώ διαφωνούμε. Στην... Το 2014 αναθεωρήθηκε με άγνωστα αποτελέσματα. Αν ζητάτε τώρα νέα αναθεώρηση χωρίς να ξέρουμε η παλιά που οδήγησε δεν είναι σωστό. Και διαφωνώ επίσης και με την αιτιολόγηση που δίνει ο εισηγητής η κυρία Κρέλ το είπε προηγουμένως, οικονομική κρίση και προσφυγική. Γιατί το συνδέεται αυτό. Όσο ε, μεγάλες και αν είναι οι επιπτώσεις και σοβαρές, δεν μπορεί να τα πάρουμε αυτά από την αλληλεγγύη μας σε θεομηνίες. Και πώς μετράτε την επίπτωση ε, ε, του προσφυγικού στη δυναμικότητα μιας περιφέρειας και άλλη γραφειοκρατία, με ποιους δείκτες θα το κάνετε αυτό. Όχι, να παραμείνει στο 1,5% γιατί αλλιώς θα μπλέξουμε με το Συμβούλιο κτλ. Πρόεδρε, να περιμένουμε τα αποτελέσματα της περασμένης αναθεώρησης. Μπορεί να έχει νόημα να τα ξαναπούμε ε, σε λίγα χρόνια. Κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ξανά ε, για να εκτιμήσουμε τι έχει γίνει. Ε, ας ελπίσουμε οι ε, περιφέρειες που πλήττονται από θεομηνίες να ενισχύονται πιο γρήγορα και όπως λέμε, λέει μια παροιμία, καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεναπεύεις ή ε, να είσαι προμηθέας παρά επιμηθέας. Ε, κυρία Βαλίνα, έχετε το λόγο. Ναι. Παρευρίσκεται κυρία Βαλίνα, εδώ είμαι λέει κυρία Βαλίνα. Sí, perdón, Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα, Πρόεδρε. Καλημέρα σα. Καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση που έκανε και για τη δουλειά του. Ε, πιστεύω πως το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα ταμείο πάρα πολύ σημαντικό για τους περισσότερους πολίτες της Ένωσης και είναι πιθανό στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ταμείο κλειδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους, αλλά και τις υπόλοιπες ε, θεομηνίες ή καταστροφές. Αλλά θα ήθελα να ενημερώσω για δύο, σύντομ, δύο μικρά λαθάκια. Από τη μια πλευρά ε, η Κομισιόν του 2014 ε, θα πρέπει να δούμε γιατί είναι λάθος και έπειτα η Επιτροπή Περιφερειών είναι του 2013 η έκθεση και όχι του 2015. Ε, θα υποβάλουμε τροπολογίες με πρόθεση να βελτιώσουμε την έκθεση ή να δώσουμε τη δική μας άποψη γιατί πιστεύουμε επιπλέον ότι είναι η στιγμή να διευρυθούν κάπως οι στόχοι αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να συμπεριλάβουν και άλλου είδους θεμηνίες όπως μπορεί να είναι οι, ανθρωπι... καταστροφές όπως είναι οι ανθρωπιστικές καταστροφές να συμπεριλαμβάνει στόχους ε, χρηματοδότησης, ε, όπως είπαμε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, θα υποβάλουμε άλλη τροπολογία ώστε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το σύστημα οικονομικών κριτηρίων ε, και επιπέδων, μάλλον κατοφλίων για την πρόσβαση στα κατόφλια, έτσι ώστε οι πιο ευάλωτες και οι πιο φτωχές περιοχές της Ένωσης να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια, ε, να έχουμε ένα σταδιακό κείμενο όπου οι πιο πλούσιες χώρες και περιφέρειες ε, να έχουν πιο ψηλά κατόφλια από ότι οι φτωχότερες. Αυτό το θέμα της σταδιακότητας, της προοδευτικότητας ε, χρησιμοποιείται εξάλλου και στα, από Υπουργεία Οικονομικών των περισσότερων κρατών μελών ήδη. Δεν έχει αλλάξει η δομή αυτού του ταμείου από τότε που δημιουργήθηκε το 2002, ενώ δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν σε περισσότερες αλλαγές και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι το, το, το, κονδύλι που προβλέπεται για το Ταμείο θα έπρεπε να αυξηθεί. Επίσης θα υποβάλουμε μια τροπολογία όσον αφορά τον γεωγραφικό ορισμό των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές. Και τέλος, ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πολιτικές ισότητας φύλου και δικαιωμάτων της γυναίκας ως κριτήριο επιλεξιμότητας των αιτήσεων. Οι γυναίκες γνωρίζουμε ότι είναι μια από τις ομάδες που ε, ε, πλήττονται περισσότερο από τις καταστροφές κάθε είδους και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διαπιστώνεται σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις και διάφορους διαπιστωθεί από διάφορους οργανισμούς, από τον ΟΗΕ, την Διεθνή Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Καταστροφών και που λέει ότι η προοπτική του φύλου θα πρέπει να εντάσσεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλες τις προβλέψεις και όλα τα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ε, κάνουν προϋπολογισμό, προϋπολογισμό του κινδύνου, και εκτιμήσεις. Επίσης, στη Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι οι γυναίκες χάνουν πολύ περισσότερο τη ζωή τους στη διάρκεια φυσικών καταστροφών από ότι οι άνδρες. Η συμπερίληψη του θέματος του φύλου στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό πριν ε, για την αντιμετώπιση καταστροφών μπορεί να σώσει πολλές ζωές. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή, πιστεύω, για να μπορέσουμε και εμείς να εντάξουμε άλλες αποστολές μέσα σε αυτό το ταμείο. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω πως έτσι θα ε, υπάρξει μια πραγματική σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και με την ευκαιρία να σας ευχηθώ και καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Και σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος είναι ο σκιώδης συζητητής κύριος Ρόπε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κίκο για, για την, ε, ε, την, ε, το σχέδιο έκθεσής του. Το Ταμείο αλληλεγγύη έχει ευγενεί στόχου να παρέχει γρήγορη βοήθεια, ταχεία βοήθεια στα κράτη-μέλη και στι περιφερειέ που έχουν υποφέρει από φυσικέ καταστροφέ. Η έκθεση αυτή απογράφει αυτέ τι δράσει, όμω υπάρχουν προβλήματα και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Είναι παράξενο που συζητάμε αυτή την έκθεση για τι δραστηριότητες του 2014 στα μέσα του 2016. Κάτι άλλο. Χαμηλό αριθμό αιτήσεων. Νομίζω πως η έκθεση, μάλλον ο εισηγητή θα μπορούσε αυτό να το τονίσει. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή γιατί, σε τι οφείλονται οι καθυστερήσει διότι δεν υπάρχουν εδώ εξηγήσει, δεν δίνονται εξηγήσει στην έκθεση της επιτροπή. Ε, στην έκθεση για το 2014 βλέπουμε ότι σε διάφορες περιπτώσεις, για παράδειγμα για την Σλοβενία, η ταχεία βοήθεια δόθηκε, καταβλήθηκε ένα χρόνο μετά από την υποβολή του αιτήματος. Πώς μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτό το ταμείο είναι ένα ταμείο γρήγορης ε, ανταπόκρισης. Γιατί η Κομισιόν σε αυτή την έκθεση δεν μας εξήγησε γιατί παίρνει περισσότερο από ένα χρόνο να δοθεί αυτή η γρήγορη ε, απάντηση και ανταπόκριση. Είμαι σίγουρη ότι, σίγουρος ότι η Κομισιόν θα μας εξηγήσει σε τι οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις, καθώς και τι μέτρα λαμβάνονται για να μειωθεί ο χρόνος απάντησης. Ε, ακόμα ένα πρόβλημα που διαπιστώνουμε είναι ότι... το κράτη-μέλη επιβαρύνονται με 10% ε, αναπόφευκτες δαπάνες. Τι είναι αυτά τα έξοδα. Διάφορα, γραφειοκρατικά, διαδικαστικά. Όταν ε, πρέπει, ε, παίρνει κανείς ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο κόσμος που δίνει αυτή τη βοήθεια να είναι βέβαιος πριν λάβει την απόφαση για χορήγηση της βοήθειας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο λόγο για πρόληψη και για προσαρμογές στις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Και αυτά να είναι η προτεραιότητά μας. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο που έχει ε, μιλήσει και για τα διαρθρωτικά ταμεία και την ευελιξία των δημοσιο... χρηματοδοτικών μέσων ε, που έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης ε, των κονδυλίων και έτσι να μπορέσουμε να αντιδράσουμε καλύτερα στις ανάγκες των ανθρώπων. Μάλιστα, συνεχίζουμε τώρα με τους συναδέλφους που ζήτησαν τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, το Ταμείο Λιλεγγύης το έχουμε ξανασυζητήσει. Θυμάμαι ότι ότι ε, ο αντιπρόεδρος, ε, ο αντιδήμαρχος μάλλον και ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής ήρθε μάλιστα στη χώρα μας όταν έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή οι πλημμύρες ε, και τότε μπορέσαμε να έχουμε πραγματικά βοήθεια, λάβαμε βοήθεια νομική, λάβαμε χρήματα και ευχαριστώ όλους διτρούς γιατί μας έφτασε μάλιστα πριν να μπούμε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ταμείο της Αλληλεγγύης να βοηθά γρήγορα. Και γι' αυτό και ευχαριστώ και τον εισηγητή που το λέει, γιατί στην ε, περίπτωση καταστροφής, ε, αν, δίνονται, αν δοθούν χρήματα γρήγορα, ε, πιάνουν διπλά τόπο. Ε, άρα λοιπόν δεν πρέπει Εντάξει, ναι, υπάρχουν κανόνες, δεν λέω, το κατανοούμε αυτό, χρειάζεται και αυστηρός έλεγχος. Όμως η εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε αυτή την περίπτωση θα ε, αυξανόταν αν μόνο ένα όργανο ήταν υπεύθυνο για να παρέμβει στην έγκριση της επιχορήγησης. Αν και οι τρεις πρέπει να εγκρίνουν, ε, ε, τότε η ταχύτητα ακυρώνεται και μειώνεται πολύ. Εδώ η ταχύτητα παίζει ρόλο. Το 2016 δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε νέους κανόνες, γιατί υπήρξε ήδη μια μεταρρύθμιση. Όμως πρέπει να πούμε σε τι κατεύθυνση θέλουμε να πάμε με το Κοινοβούλιο, γιατί ακριβώς το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να αντιπροσωπεύσει για τους Ευρωπαίους πολίτες την απτή βοήθεια όταν βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα όσα είπε η συνάδελφος για τον ευάλωτο χαρακτήρα, την ευάλωτη ομάδα των γυναικών που πολλές φορές κινδυνεύουν και από θάνατο άμεσο. Δεν το ήξερα. Η έκθεση δεν λέει τίποτα γι' αυτά. Ίσως λοιπόν θα, καλό θα ήταν να ενταχθεί αυτή η πτυχή του φίλου στην έκθεση, όπως είπε και η συνάδελφος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το μας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι αποτελεσματικό και σημαντικό εργαλείο που ιδρύθηκε το 2002 για την αλληλεγγύη προς περιοχές που πλήττονταν από φυσικές καταστροφές με τόσο σοβαρές πλημμύρες στην κεντρική ε, Ευρώπη. Αυτό το Ταμείο θα έχει σημαντικότατο ρόλο στο μέλλον για τις φυσικές καταστροφές και είναι ένα από τα βασικότερα σύμβολα αλληλεγγύης ε, όταν συντρέχει ανάγκη και γι' αυτό θα πρέπει να πλουστευτεί η διαδικασία ούτως ώστε να καταβάλλονται τα χρήματα αμέσως μετά την καταστροφή όταν υπάρχει αναγκή όπως ε, το 2013 στη Σλαβωνία στην ε, Κροατία όπως είπε και ο εισηγητής μας ο κύριος Τσίκο ε, Είχαμε τρόφιμα και ρούχα την επόμενη ημέρα, αλλά στέγη ικανοποιητική δεν είχαν οι άνθρωποι για πολλές μέρες. Επιδιορθώθηκαν τελικά οι ζημιές, αλλά τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις έμειναν όπως ήταν. Ε, δύο χρόνια μετά ε, έχετε τα κτίρια, έχετε ε, τα σπίτια, αλλά έφυγαν οι άνθρωποι Πήγανε στην Αυστραλία, πήγανε εκεί πέρα που μπορούσαν να δουλέψουν. Γιατί ξαναλέω τα εργοστάσια δεν τα ξαναφτιάξαν. Ευχαριστούμε. Ναι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις καλές του ιδέες. Ε, να σας πω πόσο σημαντικό είναι για μας το Ταμείο Λιλεγγύης. Ξέρετε ότι κατάγομαι από τις Αντίλες. Ε, δεν ξέρω αν έχετε πάει πρόσφατα. Σε 10 χρόνια ζήσαμε τρεις κυκλώνες με ε, ανέμους ε, θελώδης 300 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα και μεγάλα ελλείμματα και μας χρειάζεται πάρα πολύ αυτό το Ταμείο Λιλεγγύης. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος συγητής επιμένει πάρα πολύ στο θέμα της πρόληψης. Καλύτερη πρόληψη παρά η θεραπεία, πάντα. Και θα πρέπει να κινητοποιείται πολύ πιο γρήγορα αυτό το Ταμείο. τα ξέρουμε αυτά. Όταν περάσει μια θεομηνία δεν μπορείς να περιμένεις μήνες ολόκληρους για να αποζημιωθείς. Υπάρχουν προβλήματα ε, για ε, το πληθυσμό των αντιλών που έτσι και αλλιώς είναι σε πολύ μειονεκτική θέση. Αυτά. Ευχαριστώ. Πάντως το κείμενο είναι πολύ καλό. Θα κάνουμε και εμείς τροπολογίες. Ευχαριστώ. Άλλος, ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για την προσπάθειά του και την αξιολόγηση ε, για το τι συμβαίνει πραγματικά στην πράξη. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, οι πολίτες περιμένουν να δρούμε ταχύτερα και από την άλλη να ελέγχονται και τα πράγματα ανάλογα με το επίπεδο, την κλίμακα της θεομηνίας και κατά πόσο ε, αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό του επ της χώρας ή της περιφέρειας. Υπάρχουν κάποιες θεομηνίες ε, στις οποίες ανέφερε και ο κ. Φαν Μίλτενμπουργκ που ε, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Και αν κατεβάσουμε το κατόφλι, το κατώτατο όριο, τότε ε, μπορεί αυτό το ποσοστό να είναι πολύ μεγάλο. Ακούω στην Ολλανδία ότι στο Νότο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαλάζει, που είναι περίπου όσο αυτό το μπουκαλάκι το νερό. Ε, και έχει παραλύσει ε, μια ολόκληρη περιοχή. Όταν πέφτει τέτοιο χαλάζι σαν το μπουκαλάκι του νερού που σας δείχνω, τι να κάνεις. Και μετά σου λένε, αλλά τα όρια είναι τόσο ψηλά του ΕΠ που δεν μας κατατάσσουν σε χαλαζόπληκτη περιοχή, ας πούμε. Ως χαλαζόπληκτη. Και σου λέει υπάρχουν τα ταμεία συνοχή και πήγαινε βρέστα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθάει τους πολίτες που περιμένουν αυτή τη βοήθεια. Και όσο πιο συγκεκριμένο είσαι τόσο καλύτερα. Δεν λέω να ανατραπεί όλο το σύστημα όπως έχει σήμερα, αλλά μήπως να σκεφτούμε μια πιο στενή διαφοροποίηση. Ξέρω ότι δεν είναι νομοθετικό το θέμα, να βρούμε μια διατύπωση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, no more Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Να ακούσουμε τον κύριο Βάχτερ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ridge από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόφερα σωστά. Πολύ ωραία. Ιωάννης Βάχτερ λέγομαι από τη DG Radio. Ε, είμαι υπεύθυνο για το Ταμείο Ελληνικής καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή και όπως είπα και την περασμένη φορά θα το επαναλάβω Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους ιδιαίτερως στην Επιτροπή σας και την Επιτροπή ε, ε, των Προϋπολογισμών για την υποστήριξη προς το Ταμείο Αλληλεγγύης. Σίγουρα ε, ε, υπάρχουν ατέλειες ακόμη στο Ταμείο. Σίγουρα δεν εκπληρώνει όλες τις προσδοκίες που υπάρχουν εδώ στο Κοινοβούλιο και στις πληγήσεις περιοχές. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους μετά από φυσικές καταστροφές και είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Για 24 χώρες, κυρίως κράτη-μέλη ε, και κάποιες υποψήφιες χώρες, κινητοποιήθηκε το Ταμείο για 71 φυσικές καταστροφές και από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί 3,8 δις ευρώ. Η αναθεώρηση του 2014 επέφερε πολύ σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του Ταμείου και ρυθμίστηκαν διάφορα ζητήματα που και πάλι θέσατε εδώ σήμερα και αναφέρθηκαν και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου όταν εξέτασαν το σεισμό στο Αμπρούτσο ε, το 2008. Μετά τη μεταρρύθμι στο 14, λοιπόν, καλό θα ήταν να κρίνουμε την τρέχουσα λειτουργία του Ταμείου δυνάμεων των ε, ε, τωρινών διατάξεων. Ευτυχώς, και το τονίζω ευτυχώς το 2014 και μετά δεν είχαμε τόσο πολλές φυσικές καταστροφές, είναι απρόβλεπτα φαινόμενα. Κάποιες χρονιές έχουμε πολλές, άλλες ε, λίγες από το 2014 και μετά δεν σημειώθηκαν πάρα πολλέ φυσικέ καταστροφές και ως εκ τούτου είναι ενδεχομένως λίγο πρόωρο να κρίνουμε τώρα αν οι νέε διατάξει είναι στο ύψος των ε, προσδοκιών μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν ε, παρόλα αυτά σαφείς ενδείξεις ότι είναι απλούστερο ε, πιο ξεκάθαρο και με μεγαλύτερη δυνατότητα απόκριση στο Ταμείο Αλληλεγγύης ε, μετά τη μεταρρύθμιση. Προκαταβολές, ε, παραδείγματο χάρη, σε σχέση με αυτά που επιτρέπει πλέον ο προπολογισμός από το 2015 και μετά έγιναν και έτσι μπόρεσαν να λάβουν τα χρήματα οι πληγήσεις περιοχές. Και το σημαντικότερο είναι τα κριτήρια για τις ε, περιφερειακές ε, καταστροφές, ε, το αντικείμενο δηλαδή των σοβαρότερων επικρίσεων και που είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχουν βελτιωθεί και με τα νέα κριτήρια καμία φυσική καταστροφή δεν απορρίψαμε. Ε, σε περιφερειακό επίπεδο στο παρελθόν, επειδή δεν ήταν ξεκάθαρες διατάξεις, δύο τρίτα των ετοιμάτων ε, ε, από, στο περιφερειακό επίπεδο έπρεπε να απορριφθούν και καταλαβαίνετε την απογοήτευση αυτών που είχαν υποβάλει το αίτημα και δεν μπορούσαν να λάβουν τη συνδρομή που χρειάζονταν. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί με τις νέες διατάξεις να ελέγχει και την εφαρμογή. Την απορρόφηση των κονδυλίων πολύ στενότερα σε σχέση με το παρελθόν και να διαπιστώνει αν ε, υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες. Ε, ταχύτερα δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε αυτό τον έλεγχο. Παραδοσιακά καθυστερούσε η αξιολόγηση Φυσικά οι προϊόντες καταστροφές είναι η προτεραιότητα. Η εφαρμογή, ο έλεγχος εφαρμογής είναι κάτι απαραίτητο για λόγους αφήνειας, διαφάνειας κτλ. Αλλά ε, είναι δευτερεύοντα σε σχέση με τις ε, τρέχουσες καταστροφές. Σε κάθε περίπτωση ε, έχουμε βελτιώσει τις επιδόσεις μας σε σχέση με το παρελθόν. Α θυμηθούμε επίσης το, τη, τη, τη λογική. Γιατί ιδρύθηκε αυτό το το 2002. και παρέμεινε μετά την ε, μεταρρύθμιση του 2014 παρά τις επικρίσεις. Γιατί, όταν πλήττονται από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές τα κράτη-μέλη, όχι από όλες, αλλά στις περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη και κάποιες υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες αγωνίζονται, ε, μάχονται να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστροφές ε, τους προσφέρουμε βοήθεια στο μέτρο των πόρων που έχουμε. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, όσο και αν το θέλαμε αυτό. Υπάρχουν όρια. Τα όρια αυτά ορίζονται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μειώθηκε κατά το ίμιση η πρικοδότηση του Ταμείου στο τωρινό πολιετές, στα 500 εκατομμύρια από το 1 δις. Επίσης, ε, ένδειξη αλληλεγγύη αυτό είναι ένα ζητούμενο για την οικονομική στήριξη, δηλαδή για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικέ συνέπειες ε, των καταστροφών βάση καταστατικού δεν είναι εργαλείο κατεπίγουσας βοήθειας δυστυχώς το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ε, υπάρχουν άλλα εργαλεία γι' αυτό, από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΟ παραδείγματος χάρη. Αυτά τα μέσα επιτρέπουν στην Ένωση να βοηθήσουν με άμεση απόκριση όταν ε, συμβαίνει μια φυσική καταστροφή σε διάστημα ημερών ή και ωρών. Στέλνουν φάρμακα, αεροπλάνα και το, και το καθεξής αλληλεγγύης ε, βάση καταστατικού ξαναλέω δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Καλύπτει άλλε ανάγκες. Υπάρχουν καθυστερήσεις ε, κάποιες αδικαιολόγητες όντως. Υπενθυμίζω όμως πως δεν μπορεί να ενεργοποιήσει εξιδίας πρωτοβουλία στο Ταμείο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να περιμένουμε το αίτημα. 12 εβδομάδες είναι το αίτημα. Τρεις μήνες περνάνε οπωσδήποτε πριν αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Και πρέπει να μεταφραστεί και το αίτημα. Γιατί δεν παίρνουμε μόνο από αγγλόφωνες και γαλλόφωνες περιοχές αιτήματα, από Ελλάδα, από Εστονία. Και για τη μετάφραση θέλουμε χρόνο. Ε, ο φορολογούμενος δεν απαιτεί βάσει των διατάξεων να ελέγχουμε το παραδεκτό των ετοιμάτων. Επίσης δεν τα έχουμε τα χρήματα έτοιμα ζεστά να περιμένουν. Ε, είναι εκτός προϋπολογισμού, όπως ξέρετε, η χρηματοδότηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να δώσουν ε, μέσω τρο, διαδικασίας ε, τροποποιητικού σχεδίου του προϋπολογισμού να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ε, για να απελευθερωθούν τα κονδύλια. Οχτώ εβδομάδες είναι η διαδικασία ελέγχου για τα κονδύλια για να εκταμιευθούν. Καταλαβαίνετε, τρεις μήνες θέλουμε, λυπούμεθα. Θα θέλαμε να αντιδρούμε ταχύτερα αλλά αυτό είναι και ένα από του βασικού λόγου που δεν αδυνατούμε να ε, κινηθούμε ταχύτερα. Συμπληρωματικότητα με άλλα ε, μέσα και εργαλεία. Το θέσατε και αυτό. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνουμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια οι πόροι στα ε, επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία, στα διαρθρωτικά για την πρόληψη ε, χρησιμοποιούνται και είναι συμπληρωματικά σε σχέση με το φτωχό Ταμείο Αλληλεγγύης, 500 εκατομμύρια το χρόνο, σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για την πρόληψη και βάσει του τωρινού κανονισμού δεν προβλέπεται παρέμβαση και διαφορετικού τύπου καταστάσεις, ε, όχι φυσική καταστροφή, π.χ. ανθρωπιστική καταστροφή, προσφυγική, οικονομική κρίση. Το έχουμε συζητήσει αυτό. με την ευκαιρία της τελευταίας μεταρρύθμισης, ε, δυστυχώς ε, εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Και εξυπακούεται ότι εμείς ε, ευθυγραμμιζόμαστε με το πεδίο εφαρμογής. Ξαναλέω, όπως και στην αρχή της παρέμβασής μου, σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε τις διοικητικές ε, βελτιώσεις που χρειάζονται για να επισπεύσουμε τη διαδικασία, να αυξήσουμε τη διαφάνεια και πάλι σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την εξαντλητική ε, παρουσίαση. Και... Κύριε Τσίκου, ε, να κλείνουμε σιγά σιγά. Κύριε Τσίκου, να κλείσουμε. Ε, ναι, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν ε, σημαντικά σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και να ευχαριστήσω και την Κομισιόν που έδειξε τη διάθεσή της να βελτιώσει περισσότερο αυτές οι διαδικασίες που θέσαμε στην, παραθέσαμε στην έκθεση που ξεκινούν από την αργοπορία, την έλλειψη συνεργασίας αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια. 18 Ιουλίου με την κατάθεση των τροπολογιών θα κατανοήσουμε ακριβώς τι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στην έκθεση και να επίσης να σας ευχηθώ και εγώ καλές διακοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λεπτάκια δώστε μου για να κλείσουμε τη σημερινή μέρη σε διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Συνεδρίασαν εχθές το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Κυκλοφόρησαν με mail, σας εστάλησαν εχθές το βράδυ οι αποφάσεις τους. Τις δέχεστε? Yes. Ναι. Από ό,τι φαίνεται εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των συντονιστών. Διάφορα. Έχουμε τίποτα στα διάφορα. Όχι. Κύριε Βανίστερο, Ρόι, δεν έχετε κανένα διάφορο. Τι πάθατε. Είστε για διακοπές έτοιμος. Ωραία. Ε, θυμίζω την προσεχή συνεδρίασή μας είναι στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα 5η από τις 9 το πρωί ε, και όλη μέρα. Ευχαριστώ και τους Δερμηνείς. Ευχαριστούμε. Και επίσης εύχομαι σε όλους σας καλές διακοπές με ήλιο, με ηρεμία να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά και να εμπνευστείτε. Για να είστε έτοιμοι για τη σκληρή δουλειά που μας περιμένει το φθινόπωρο με το καλό. Λέξη συνεδρίασης. Καλό σας καλοκαίρι.